Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανάπτυξης, διότι εκ νέου επελήφθη αυτού του ζητήματος και να επαναβεβαιώσω την τη στήριξή της στην καταπολέμηση αυτού του μεγά έργου, το οποίο θα έχει και θα επιφέρει τεράστιες περιβαλλοντικές ζημίες και καταστροφικές επιπτώσεις επί του τοπικού πληθυσμού. Όπως ε, σωστά υπενθύμησε η πρόεδρος μας, επιτόπου δίνουν μάχη και πληρώνουν μέσα με τη ζωή τους τον αγώνα που δίνουν για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της βιοπικιλότητος. Το γνωρίζετε αυτό ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουμε κινητοποιηθεί για να γίνει ακουστή και να ακουστεί η φωνή τους έχοντας με γραπτό ερώτημα θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 έχοντας προσωπικώς προειδοποιήσει την κυρία Άστον το Μάιο του 2010 Έχοντα φροντίσει να συμπεριλάβουμε αυτή μα την ανησυχία στο κοινοβουλευτικό μα έργο, στι δύο εκθέσει, παραδείγματο χάρη οι οποίε αναφέρθηκαν προηγουμένω, όσον αφορά την πρόσβαση, την παγκόσμια πρόσβαση στην ενέργεια στι αναπτυσσόμενε χώρε, ή ακόμη και στην έκθεση τη σχετική με τι υποδομές αν θέλετε και τις, τα φράγματα και ω συντονίστρια τη ομάδα των Πρασίνων χρησιμοποίησα τα διάφορα θεσμικά μέσα που είχα στη διάθεσή μου και τα μέσα που είχα στη διάθεσή μου σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ευαισθητοποιήσω στη σημασία του ζητήματος αυτού. Επειδή αυτό το μέγα έργο είναι αντίθετο προς το σύνταγμα της χώρας. Πράγμα το οποίο αναγνωρίστηκε εξάλλου και από τα όργανα της ε, βραζιλιανής δικαιοσύνης. Διότι σύμφωνα με το σύνταγμα της Βραζιλίας θα έπρεπε προηγουμένω να υπάρξει διαβούλευση με τους αυτόχρονους πληθυσμούς. Αυτό βεβαίως δεν παρεμπόδισε την κατασκευή η οποία ξεκίνησε τον 28 Αυγούστου που μας πέρασε. Και διότι στο επίκεντρο αυτής της μάχης μεταξύ της κυβερνήσεως και των ντόπιων πληθυσμών είναι η επιλογή του τρόπου ενεργειακής ανάπτυξης. Και υπενθυμίζω ότι το κόστος του φράγματος ανέρχεται γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, 10 δις ευρώ, για μια πρόβλεψη 11.233 ΜΒ ισχύω, αλλά μόνο 4.500 θα εξασφαλίζονται κατά τους 6 μήνες του έτους και μόνο 13% θα χρησιμοποιείται σε τοπικός, ενώ το 30% θα μεταπολείται στο εξωτερικό. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δεχθεί, ερώτω, ή και το, χειρότερο μπορεί να συμμετάσχει έμεσα σε αυτές τις αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών. Καταστροφή του Αμαζονίου. Πνεύμονας για όλους μας και για καθαρά οικονομικούς λόγους μπορούμε να το δεχτούμε αυτό και να το στηρίξουμε. Αν δεν δεχτούμε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, τότε οι δικέ μα επιχειρήσει δεν πρέπει και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην κατασκευή αυτού του έργου. Γνωρίζουμε όλοι μα εδώ ότι οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει εμπλέκονται και συμμετέχουν. Επομένω, το ερώτημά μου είναι απλούστατο. Τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλει να κάνει προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κυβέρνηση τη Βραζιλίας και επίση και κυρίω τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο ζήτημα αυτό και να φροντίσει έτσι τουλάχιστον οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές εταιρείες να μην συμμετάσχουν σε αυτή την καταστροφή της βιοπικιλότητος και αυτό αγνοώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και των αυτοκτόνων πληθυσμών. Και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκπροσωπείται από τον κύριο Νίκολας Χάνλεϊ και τον κύριο Ατιέν Κογιέτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριοι και κυρίες Ευρωβουλευτές, όπως θα γνωρίζετε, πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο σε δύο φορές έχει απασχολήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γραπτές ερωτήσεις προς την κυρία Άστον, την Επίτροπο Άστον και στις οποίε δόθηκαν απαντήσει. Συμπληρώνω όμω αυτέ τι απαντήσει με συρωματικέ πληροφορίε και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία τέθησαν σήμερα. Θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω Λέγοντά σα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή ζητήματα που έχουν σχέση με την κατασκευή αυτού του έργου. Αλλά όπω υπόθηκε σε προηγούμενε απαντήσει από την Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κατασκευή αυτού του φράγματο αποτελεί αν θέλετε μια εθνική προσπάθεια και η εκτέλεσή του είναι ζήτημα εθνική κυριαρχία για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άμεσο δικαίωμα και δεν μπορεί να επέμβει. Θα ήθελα επίση να σε ενημερώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, έχει τακτικού διαλόγου με την κυβέρνηση τη Βραζιλία πάνω σε περιβαλλοντική φύσεω θέματα, όπω επίση και ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό ο τελευταίο διάλογο περιλαμβάνει και συζητήσει για θέματα που έχουν σχέση με του ε, πληθυσμού, του ντόπιου πληθυσμού. Όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, γνωρίζουμε την έκθεση στην οποία αναφέρθηκε και η, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει υπόψη τη εργασία τη Διεθνού Επιτροπή για τα Φράγματα που όπω είπατε Πρόεδρε έχει θέσει θεμελιώδη φύσεω ερωτήματα όσον αφορά τα φράγματα και τη συνεισφορά του και τη συμβολή του στην ε, ενέργεια κτλ. κτλ. Ο, όλα αυτά είναι συστάσεις από την Επιτροπή αυτή προς τα μέλη των ΗΕ, ζητώντα ζητώντας τους να λάβουν υπόψη τους τα ζητήματα των κερδών που θα μπορούσαν να προκύψουν από την κατασκευή τέτοιου είδους φραγμάτων. Αλλά όπω σας λέω αυτό πρόκειται για επιμέρους αποφάσει κυρίαρχων κυβερνήσεων και κρατών. Και στο πλαίσιο τη στρατηγικής εταιρική σχέση για το περιβάλλον που ξεκίνησε το 2007 με τη Βραζιλία και οι περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα συζητώνται τακτικά. Για να γίνει αυτή η εταιρική σχέση επιχειρησιακή και λειτουργική και για να υπάρξει αυτός ο διάλογος για το περιβάλλον και το κλίμα. Το φράγμα του Μπελομόντε είναι ένα εθνικό έργο και σε απάντηση ερωτήσεων που θέσατε, θα ήθελα να σας θυμίσω τις απαντήσεις που λάβατε προηγουμένως. Ότι δεν υπάρχει κοινοτική ευρωπαϊκή ενωσιακή χρηματοδότηση. Ούτε πηγές, ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή από τα αναπτυξιακά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επομένως, η κατασκευή αυτού του φράγματος στη Βραζιλία είναι εσωτερικό ζήτημα. Τη Βραζιλία δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα, δεν μπορεί να παρέμβει. Αλλά στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δράσεων συνεργασία την προστασία και την διατήρηση στην περιοχή του φράγματο. Και αυτό αναφέρθηκε και από εσά, Πρόεδρε. Projects, έργα δηλαδή, τα οποία βοηθούμε εμεί, βοηθούμε το, το κράτο Βραζιλία προκειμένου να έχουμε αηφόρο ανάπτυξη των δασών και διαχείριση αυτών, στην οποία θα συμμετέχουν βεβαίω και οι ντόπιοι πληθυσμοί, με μια βιώσιμη εκμετάλλευση χωρί απώλεια δασών και δάσου. Όσον αφορά το ζήτημα τώρα των αυτοκτόνων πληθυσμών, είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η Βραζιλινή κυβέρνηση στο 1992, μάλιστα, θέσπισε εθνικά μέτρα, προκειμένου να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των γηγενών πληθυσμών. Και η Βραζιλία, όπως γνωρίζετε, και την Διεθνή Σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού εργασία για τους ε, αυτόχθονες και ε, ηθαγενεί πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου με τη Βραζιλία στις 10 Σεπτεμβρίου φέτος, τα δικαιώματα των αυτοκτόνων πληθυσμών. Υπό το φως προσφάτων ανακοινώσουν Περτολία 2003 που εξέδωσε η Γενική Εισαγγελία της Βραζιλίας για αναφορικά με το μέλλον της οριοθέτησης των περιοχών που ανήκουν σε αυτόχρονους πληθυσμούς, όπως και το ζήτημα αυτού του φράγματος, συζητήθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει και επισημαίνει ότι η Βραζιλία και άλλες αμερικανικές χώρες θα πρέπει να στηρίξουν έτσι ώστε να διατηρηθεί η ανεξαρτησία και να προστατευτεί το σύστημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αμερική. Και οποιαδήποτε αποδυνάμωση θα πρέπει να αποφευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα έθεσε τέτοιε περιπτώσεις για ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εκφοβίστηκαν ή δολοφονήθηκαν και ενημέρωσε ότι η πρόθεση και η προαγωγή και η προστασία βρίσκεται στην καρδιά της ε, Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναφέρθηκε και το φράγμα του Μπελομόντε και ότι οι διαβουλεύσεις που γίνονται και συνεχώ από τότε που ξεκίνησε ο σχεδιασμό προ δεκαετία και αποτέλεσαν μια περίπλοκη διαδικασία. Αρνήθηκαν οτιδήποτε επαφή με τον έξω κόσμο και οι διαβουλεύσεις συνδέθηκαν με το πρόγραμμα Ενέργεια για όλου και στι πλέον απομακρυσμένε περιοχέ του Αμαζονίου. Η Βραζιλία επεσήμανε και τόνισε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να συντονιστούν τα συμφέροντα όλων των αυτοκτόνων πληθυσμών και εκείνων που χρειάζονται την ενέργεια. Η Βραζιλία είχε την εκτελεστική γραμματεία τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επίση. με την οποία το ζήτημα των μέτρων προφύλαξη συζητήθηκε και ετέθη. Θα πρέπει επίση να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργώ παρακολουθεί επί σειρά ετών τα δικαιώματα των αυτοκτόνων και γηγενών πληθυσμών μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων και ελέγχει τις γραμμές του προπολογισμού. Και η, η πρωτοβουλία της Ένωσης για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα χρηματοδούμενα αυτά projects έχουν στόχο να ενδυναμώσουν και να ενισχύσουν τους γενείς πληθυσμού προκειμένου να μπορέσουν να αξιώσουν και να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους στην γη και στην χρήση γης και στην αξιοποίηση αυτής. Κάποια από αυτά τα projects δίνουν, ε, προσφέρουν προστασία στους γενείς πληθυσμούς και από μη κυβερνητικό οργανισμό της Βραζιλίας αποσκοπεί και έχει σαν στόχο τους γηγενείς πληθυσμού στις ποτάμιες ε, λεκάνες που επηρεάζονται και θα επηρεαστούν από το φράγμα του Μπελομόντε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα δικαιώματα των αυτοκτόνων πληθυσμών και έχει στηρίξει μια σειρά έργων που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τους γηγενείς πληθυσμού προκειμένου να μπορέσουν να αξιώσουν και να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους μέσω μη κυβερνητικών οργανισμών της Βραζιλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτή είναι σε ενισχύ επαφή με τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών τη Βραζιλία και εκπροσώπου των γηγενών αυτοκτόνων πληθυσμών. Τώρα έρχομαι στο ερώτημα το οποίο έθεσε η κυρία Γκρέις. Θέσατε το ερώτημα του κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα ρόλο που μπορεί να παίξει, επηρεάζοντα τι αποφάσει τη βραδινή κυβέρνηση. Οφείλω να ομολογήσω ότι η δήλωση που σα διάβασα είναι μια δήλωση την οποία ετοιμάσαμε από κοινού οι διάφορε υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση του θέματο αυτού από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεπώ, δεν έχει λάβει θέση επί του θέματο αυτού. Και όπω υπόθηκε δύο φορέ στι απάντηση γραπτών ερωτήσεων, από την Αντιπρόεδρο Άστον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι αυτή η απόφαση σχετική με το φράγμα είναι απόφαση τη βραζιλινή κυβέρνηση κυριάρχου κράτου για την οποία δεν υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα, ενωσιακή αρμοδιότητα. Τώρα, ει απάντηση του ρωτήματο που ετέθησε σε σχέση με την θέση των πληθυσμών, δεν είμαι σε θέση και δεν μπορώ να απαντήσω ω εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά νομίζω ότι με τις γραπτές αυτές τις ερωτήσεις που θα θέσατε θα λάβετε απάντηση είτε από το Συμβούλιο των Υπουργών είτε από την Προεδρία η οποία ενεργεί για λογαριασμό του Συμβουλίου. Ζητήματα που άπτονται αποφάσεων των επιμέρους ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βραζιλία είναι θέματα για αυτές τις εταιρείες τις ίδιες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λόγο επί του θέματος αυτού. Νομοθετική ή άλλη βάση δηλαδή, για τις οποίες θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις περί επενδύσεων αυτών των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε τον Επίτροπο Πίμπαλξ. Νομίζω λοιπόν πως θα σταματήσω εδώ τη συζήτηση για το φράγμα του Μπελομόντε τις προφορικές ερωτήσεις να σας θυμίσω ότι έχετε μέχρι τις 11 Οκτωβρίου προκειμένου να καταθέσετε τροπολογίες στις προτάσεις ερωτήσεων όπως διατυπώνονται. Και θα υιοθετήσουμε το οριστικό κείμενο της ερωτήσεως ή των ερωτήσεων κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου, της δικής μας Επιτροπής εννοείται. Non, Je souhaite chaleureusement la bienvenue. Καλωσορίζω θερμότατα τον Επίτροπο Πίμπαλξ που ήρθε να συζητήσει μαζί μας για τους στόχους της ε, χιλιετίας, τους αναπτυξιακούς και πιθανά σενάρια για να προετοιμάσουμε τη μετά το 2015 εποχή, διότι δυστυχώς δεν πρόκειται το 2015 να έχουμε ε, καλύψει τους 8 στόχους που είχαμε βάλει ως ορόσημο 189 χώρες τη Βεβαίως έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι από το 2000, αλλά απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν μέχρι το 2015. Και έχουμε όλες τρία χρόνια μπροστά μα. Και οι πρόοδοι που έχουν γίνει ήταν ε, άνισες ανάλογα με τη χώρα και την περιφέρεια και ορισμένοι ε, στόχοι μας φαίνονται σήμερα άπιαστοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως είναι σταθερά προσιλωμένη σε αυτή την προσπάθεια. Ε, του χρόνου τα Ηνωμένα Έθνη θα κάνουν εκ νέου αξιολόγηση των προόδων που έχουν γίνει για τους στόχους χιλιετίες και θα προτείνουν ένα απτυξιακό πλαίσιο για τη μετά το 2015 εποχή. Τον Ιούλιο του 2012 ο Γενικός Γραμματέας του ο κ. Μπαν ανακοίνωσε ότι ο Επίτροπος κ. Πίβαλξ ορίστηκε μέλος του πάνελ υψηλού επίπεδου για την ατζέντα μετά το 2015 και στις 25 Σεπτεμβρίου ε, ήδη συμμετείχε ο κύριος Πίμπαλκ στην πρώτη συνεδρίαση του πάνελ και περιμένουμε με μεγάλη περιέργεια να ακούσουμε τα όσα διεμήφθησαν εκεί. Ξέρουμε ότι έχει αρχίσει και δημόσια ακρόαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Διαβούλευση μάλλον. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Μπίπαλξ θα ήθελα να επιμείνω στο εξή, αν επιτρέπετε. Η παγκόσμια στρατηγική για την ανάπτυξη μετά το 2015 έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικές προκλήσεις σε σχέση με αυτές που είχαμε το δεκαετία του 90 του περασμένου αιώνα. Το παγκόσμιο οικονομικό και ιδεοντολογικό και ηθικό πλαίσιο έχει αλλάξει εκ με την αλλαγή της χιλιετίας. Και τώρα ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες πραγματικότητες σε ένα νέο κόσμο. Κύριε Επίτροπε, Πίβαλ, σας δίνω μέσω στο λόγο και χρόνο έχουμε, μην ανησυχείτε. Thank you, Eva. Ευχαριστώ, Εύα. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που έχω την ευκαιρία να τόσο νωρίς στην ε, σχετική συζήτηση, έχω την ευκαιρία να παρευρεθώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Συνεργασίας και να συζητήσω τα σχετικά ζητήματα μεταξύ σας, μαζί σας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ, ο κ. Μπανκιμούν, έχει συγκαλέσει ένα πάνελ υψηλού επίπεδου για την ε, ανάπτυξη. Συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος της Λιβερίας, της Ινδονησίας, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και, προσ... και όπως βλέπετε προσπαθεί να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των αναπτυσσόμενων και των υποανάπτυξη χωρών. Ε, βλέπετε, ας πούμε, η Ινδονησία βρίσκεται κάπου ενδιαμέσως ε, μεταξύ μιας αναπτυγμένης χώρας ή μιας χώρας όπως η Κίνα. Ε, άρα μπορώ να πω ότι η σύνθεση του πάνελ συμπεριλαμβάνει 26 μέλη, ε, πρόεδρος Κέλλαρ από την Γερμανία, ο πρώην υπεύθυνο ε, αναπτυξιακής συνεργασίας από τη Γαλλία, ε, εγώ και ο Σουηδός συναδελφός μου. Συμμετέχουμε με την προσωπική μας ιδιότητα και φυσικά όταν συμμετέχει ένας Ευρωπαίος Επίτροπος σε, μια, ένα τέτοιο πάνελ. Σε κάθε περίπτωση δεν σκέφτεται μόνο ε, προσωπικά, αλλά και τι ε, επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας κάποιες προσωπικές μου σκέψεις από αυτήν την ε, συναντήση. Στο πρώτο συνάντηση μας έδωσε μια κατεύθυνση γενική ο κύριος Πανκιμούν. Όλη η διαδικασία πρέπει να είναι πλήρως ανοιχτή χρειάζομαι να καταλήξουμε σε μια έκθεση την οποία να μπορούμε να αξιοποιήσουμε το Σεπτέμβριο. Δεν ε, μας έδωσε έτσι, ε, περιοριστικούς όρους, ήταν ε, ο στόχος του να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα. Πιστεύω ότι το, η πρώτη συνάντηση ήταν κυρίως προς ανατολισμού, ήταν μια εισαγωγική συνάντηση η επόμενη στο συνάντηση στο Λονδίνο στις 31 Οκτωβρίου και 1η και 2η Νοεμβρίου. Εκεί θα συμμετάσχουν και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε, να, να συμμετάσχουν και άλλοι. Και στην παρουσίαση μου σήμερα θα μιλήσω και για την δημόσια συμβουλευτική διαδικασία που διαξήγαμε και τι αποτελέσματα έχει εκείνη. Για να πιάσουμε και τον σφιγμό. Ως Επίτροπος, τι θα ήθελα να επιτύχω. Νωρίς το επόμενο, το 2013, να έχουμε καταλήξει σε μια κοινή αντίληψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα θέλουμε να πετύχουμε μέσω από αυτή τη διαδικασία. Είναι σημαντικό να πετύχουμε μια κοινή στάση και με βάση αυτή την κοινή στάση να πάμε στο διάλογο με τους εταίρους μας. Γιατί ε, μια διαδικασία τέτοια θα μπορούσε να μας θυμίσει το προβλήματα που είχαμε στο Rio Plus, όταν κατηγορηθήκαμε ότι χάναμε χρόνο στον συντονισμό των κρατών μελών μεταξύ τους παρά με, τη με την ίδια τη διαδικασία. Γι' αυτό θα ήθελα ε, να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό που έχουμε αν συνεργαστούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 27 κράτη-μέλη. Και την περίοδο που έρχεται θα πρέπει να συνεργαστούμε και με την κοινωνία των πολιτών, ιδίω από τις ε, χώρες υπό έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια θέση, σε, μια, σε ένα κόνσεπτ, σε μια λογική που θα είναι ακριβώς αυτή που εκείνοι επιθυμούν να έχουμε κι εμείς. Θεωρώ ότι είναι χρυσή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει, να σφυριλατήσει το μέλλον μετά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Ο γενικός στόχος ήταν η εξάλληψη της φτώχειας. Αυτό ήταν και το μήνυμα από το Ρίο. Οι υποανάπτυξη χώρες σήμερα χρειάζεται να καταπολεμήσουν πρωτίστως τη φτώχεια. Και ο ρόλος μας εμείς είναι αυτός ο στόχος της καταπολέμησης της φτώχειας να γίνει με ταυτόχρονη καταπολέμηση του αποκλεισμού και με βιώσιμο τρόπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση εστιάζουμε στην καταπολέμηση της φτώχειας. τι θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε στο πλαίσιο του πάνελ επίπεδου. Πρέπει να αλλάξουμε ε, κατεύθυνση σε σχέση με το τι πετύχαμε με τους αναπτυξιακούς ε, στόχους της χιλιετίας μεταξύ τώρα και το 2015. Είναι σαφές ότι δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε όλους τους στόχους, αλλά δεν πρέπει να τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Πιστεύω ότι το 2015 είναι στο, βρίσκεται στο μέλλον. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να τους επιτύχουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, ακόμα και αν οι κάποιες προβλέψεις αυτή τη στιγμή είναι δυσμενείς. Μπορεί να τους πετύχουμε το 2020, 30, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να εργαστούμε. Προς εκείνη την κατεύθυνση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι η ατζέντα για το 2015 και μετά θα πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξη από αυτήν που έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν το, τη δεκαετία του 1990, στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και από τότε ο κόσμος έχει αλλάξει άρδιν, οικονομικά, ε, τεχνολογικά αλλά και πολιτικά και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για παράδειγμα, έχουμε δει πως μια, ένα κράτος όταν έχει καλή χρηστή διακυβέρνηση και δέχεται και μια βοήθεια με έξυπνο τρόπο, μπορεί πολύ γρήγορα από την ακραία φτώχεια να φτάσει σε επίπεδα μέσου εισοδήματος. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να προστατεύουμε και το περιβάλλον κατά την προσπάθεια μας να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Άρα η εξάλληψη της φτώχειας πρέπει να γίνει με βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε τα προβλήματα, τα περιβαλλοντικά να μην έρθουν να κυνηγήσουν τις επόμενες γενιές. Ο στόχος των αναπτυξιακών στόχων της χιλιατίας ήταν να εξαλείψουμε την ε, φτώχεια μέσα σε μια γενιά. Και αυτό ήταν αφελές. Γι' αυτό είχαν ε, διαμορφωθεί και στόχοι σχετικοί, αλλά για παράδειγμα στην εκπαίδευση μπορούμε να πούμε ότι τον πετύχαμε τον σχετικό στόχο, την εξασφάλιση της πρωτοσβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν ε, εκατομμύρια παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση τέτοια. Άρα, δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πετύχαμε αυτό που επιθυμούσαμε. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στην κατάπτυση των στόχων μας, από εδώ και πέρα, δεν ναι, συμφωνώ με τις προσεγγίσεις που λένε να μειώσουμε κατά το ίμιση, αλλά χρειάζεται, πιστεύω, να πετύχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο σε διάφορες τομείς για κάθε άνθρωπο που ζει σε αυτόν τον πλανήτη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και εσείς πρέπει να υποστηρίξετε την διαδικασία των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι δεν πετύχαμε τον έναν ή τον άλλον. Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τα απλά ζητήματα. Αλλά στα πιο περίπλοκα ζητήματα δεν τα καταφέραμε τόσο καλά. Για παράδειγμα, την υγεία των γυναικών εκεί δεν ήταν απλώς η παροχή νοσοκομιακής περίθαλψης, ήταν πιο περίπλοκο το ζήτημα. Υπάρχουν στοιχεία που, στα οποία μπορούμε να ασκήσουμε κριτική, αλλά πρέπει αυτή η κριτική να μας οδηγήσει να κάνουμε και το επόμενο βήμα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν μιλάμε για την, α, εξάλληψη της φτώχειας ως κύριο στόχο. Οι αλλαγές παγκόσμιες και οι ευκαιρίες που μας δίνει η τεχνολογία δεν θα πρέπει, μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε φιλόδοξοι στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την φτώχεια. Η MDG, η αναπτυξιακοί στόχοι της ηλετίας από μόνος τους, μόνοι τους, είναι σημαντικά θέματα που προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν, αλλά από μόνα τους αυτά δεν εξασφαλίζουν η αξιοπρεπή ζωή για όλους και πιστεύω ότι το όραμα μας για το 2030 θα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή ζωή για όλους. Το δεκαετία του 90 ήταν λογικό, βλέπαμε τους αναπτυξιακούς στόχους της γηλετίας να εστιάζονται στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Σήμερα όμως έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Πολίτες ε, σε, και σε φτωχές χώρες αλλά και σε αναπτυγμένες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φτώχειας. Και αυτούς πρέπει, σε αυτούς πρέπει να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Και οι πλούσιες χώρες μπορεί να έχουν φτωχούς πολίτες. Εδώ λοιπόν έρχεται το ζήτημα της καταπολέμησης του αποκλεισμού. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτές τις προκλήσεις μετά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, η Επιτροπή ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Πάνω από 100 ε, συμμετοχέ συνεισφορές είχαμε και ήταν σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών υποστηρίζει έντονα τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και αντιλαμβάνεται το σημαντικό τους, ε, το σημαντικό τους ρόλο. Συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δαπανίσουμε σε πολλά χρήματα για αυτούς τους στόχους, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας λένε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τους λόγους που βρίσκονται στη ρίζα της φτώχειας. Τις συγκρούσεις, την οικονομική ανάπτυξη, τη χρηστή διακυβέρνηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προστασία των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τη δημογραφική αλλαγή και την κλιματική αλλαγή. Έχοντας λοιπόν αυτά στο μυαλό, ένα πρόγραμμα για την αξιοπρεπή διαβίωση όλων θα βασιζόταν σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος, να επικυροποιήσουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, έτσι ώστε οι νέοι στόχοι να αναφέρονται στην παροχή αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους. Δηλαδή ελάχιστα όρια κάτω από τα οποία να μην βρίσκεται κανένας πολίτης στον κόσμο, κανένας άνθρωπος στον κόσμο. Συνεχίζει να είναι σαφές ότι η εξάλληψη της φτώχειας παραμένει απόλυτη προτεραιότητα. Αυτή η ας πούμε αναπτυξιακή στόχη της χιλιετίας πλας θα ε, απαιτούν οι κυβερνήσεις να τους υλοποιήσουν μέχρι το 2030 το αργότερο και στην περίπτωση των πλέον ε, φτωχών κρατών με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας και της αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας από μόνοι τους δεν ε, εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Άρα χρειάζεται επίσης να ασχοληθούμε με ζητήματα ανθρωπινών δικαιωμάτων, ισότητας, δικαιοσύνης Επίσης, δεν μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση η οποία να μην είναι βιώσιμη. Ας σκεφτούμε ότι ο πληθυσμός της γης μπορεί μέχρι το 2050 να φτάσει στα 9 δισεκατομμύρια. Θα αυξηθεί η ζήτηση κατά 50% για τροφή, για, διατροφή και κατά 40% για ενέργεια. Άρα η διάσταση της βιωσιμότητας βρίσκεται στην καρδιά της προσπάθειας της εξάλληψης της φτώχειας. Γιατί είναι σαν να κάνουμε ένα άλμα και μετά να προσγειωνόμαστε και πάλι, εάν δεν λάβουμε υπόψη μας την βιωσιμότητα. Δεν, λοιπόν, δεν υποτιμώ λοιπόν τις δυσκολίες αυτούς της ε, προσπάθειας και ιδίως μετά το Ρίο Πλασίκωση. Πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό που ονομάζω χρηστή αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Κάθε κυβέρνηση έχει υποχρεώσεις ε, έναντι των πολιτών της να αξιοποιεί με σωστό τρόπο, με χρηστό τρόπο τους φυσικούς πόρους. Είτε είναι τα δάση, είτε είναι τα ορυκτά καύσιμα, οτιδήποτε άλλο. Η χρηστή αξιοποίηση όμως συμπεριλαμβάνει και την χρηστή τη ε, αξιοποίηση των εσόδων από την αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Με τις δύο αυτές τις διαστάσεις μπορούμε να οδηγηθούμε σε σαφείς στόχους, τους οποίους κάθε πολίτης μπορεί να αντιληφθεί και να αντιληφθεί τη σχέση τους με αυτούς. Έτσι θα είχαμε ένα πλαίσιο για να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπή διαβίωση για όλους. Μπορεί να ε, ερωτηθούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ SDG και MDG. Πρέπει να δούμε εις βάθος τι θέλουμε τελικά να πετύχουμε αλλά οι δύο αυτές ομάδε στόχων συγκλίνουν, στην ίδια κατεύθυνση πηγαίνουν. Πρέπει να αποφασίσουμε που θέλουμε να φτάσουμε. Ε, αν προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τεχνητούς φραγμούς ή τεχνητές διακρίσεις μεταξύ των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας ή της συζήτησης περί βιωσιμότητας, πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. αυτά, αυτές οι δύο συζητήσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. τώρα. Θέλω να συζητήσω πώς μπορούμε... Ποια είναι η σχέση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας με το MFF. Όπως γνωρίζετε, οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας πράγματι έχουν επιτύχει πολλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σημαντικό ρόλο στην επίτευξή τους. Ε, έχει, γίνει, έχει έρθει στο προσκήνιο της πολιτικής ατζέντας η καταπολέμηση της φτώχειας και ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας έχει μειωθεί από 600 εκατομμύρια, κατά 600 εκατομμύρια από το 1990. Αλλά η πρόοδος δεν ήταν ίδια σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στην Ποσαχάρια Αφρική η θνησιμότητα των παιδιών κάτω των 5 ε, ετών συνεχίζει να είναι δύο φορές μεγαλύτερη από την αμέσως ε, λιγότερο φτωχή περιοχή. Λοιπόν, χρειάζεται να εστιάσουμε σε εκείνες τις χώρες και σε εκείνους τους τομείς που έχουν μείνει πίσω. Χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση, ε, για παράδειγμα ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την πρωτοβουλία των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Αλλά η πρωτοβουλία για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας επίσης δείχνει ότι ε, η χρηματοδότηση πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με μια έξυπνη πολιτική. Το γνωρίζω ότι αντιλαμβάνεστε τη σημασία που έχει μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας να βοηθήσουμε τις ε, χώρες εταίρους μας να επιτύχουν τους στόχους τους μέχρι το 2015 και μετά το 2015 αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι μετά το 2015 το περιβάλλον θα αλλάξει το πεδίο, την κατάσταση και το θέμα θα είναι πια η δικαιότερη κατανομή των πόρων ανάμεσα στον αναπτυγμένο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη ε, μεγάλη οικονομία, ε, παγκόσμια οικονομία, η οποία ε, δίνει στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες πρόσβαση ανεφθασμών. Συνεχίζει, συνεχίζεται, θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν αυτές τις προσπάθειες και να δείξουμε στους πολίτες και τους φορολογούμενους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα μεγάλα χρηματικά ποσά που δαπανούμε στην αναπτυξιακή συνεργασία και βοήθεια δίνουν τη μέγιστη τα μέγιστα αποτελέσματα. Σας το λέω ξεκάθαρα ότι αντιλαμβάνομαι πόσο βαριά και σημαντική είναι η ευθύνη να ε, αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα των Ευρωπαίων Φερολογούμενων Το γεγονό ότι βρισκόμαστε στο μέσο μια οικονομική κρίση είναι ένα λόγο που θα μα κάνει ακόμα περισσότερο να πρέπει να δαπανούμε αυτά τα ε, χρήματα με σοφό τρόπο, με έξυπνο τρόπο. Ήδη τα καταφέρνουμε καλά σε αυτό το τομέα. Ανεξάρτητοι οργανισμοί αναγνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό δωρητή. Η οργάνωση Publish What You Fund ε, πρόσφατα ανέδειξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους πέντε πλέον διαφανείς ε, δωρητές ε, στον κόσμο. Τους πέντε δωρητές στον κόσμο με τις καλύτερες διαδικασίες διαφάνειας και χαρά καλωσορίζω αυτά τα αποτελέσματα. Βεβαίως και μπορούμε να βελτιωθούμε. Αλλά φαίνεται ότι είμαστε ήδη σε ένα καλό επίπεδο και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Άρα και άλλες ε, χώρες άλλοι που παρέχουν βοήθεια αντιλαμβάνονται την προστιθέμενη αξία που φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναπτυξιακή συνεργασία. και θα ήθελα αυτό να συνεχιστεί και τα επόμενα 7 χρόνια στο πλαίσιο του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Για μένα το να βρισκόμαστε ανάμεσα στους καλύτερους στον κόσμο δεν μου αρκεί. Εργαζόμαστε πολύ ε, σκληρά για να ετοιμάσουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο του προπολογισμού για το ε, να εστιάσουμε σε ορισμένες προτεραιότητες, συγκεκριμένες προτεραιότητες, για να γνωρίζουμε ακριβώς τι προσπαθούμε να πετύχουμε τα επόμενα αυτά χρόνια. Την κοινωνική προστασία, την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς επίσης και την, ε, τη διάρκεια. Δηλαδή, έχουμε αντιληφθεί ότι από τη στιγμή που δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να τον λαμβάνει υπόψη της και η αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει να προσπαθούμε να δημιουργούμε λύσεις που διαρκούν σε μια ε, χώρα έτσι ώστε να μην χρειάζεται συνέχεια ανθρωπιστική βοήθεια μια χώρα. Μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας να λύσει το πρόβλημά της πιο μακροπρόθεσμα. Ε, πιστεύω ότι το καλύτερη κριτική είναι η υποκοδομητική κριτική αυτή που λέει ότι αργούμε πολύ, ότι οι διαδικασίε θα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορες. Και επίσης η προβλεψιμότητα της βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει οι κανόνες και οι συμφωνίες που κάνουμε με τους εταίρους μας να είναι σαφέστατες, δηλαδή από τη στιγμή που θα τηρηθεί συμφωνία θα υπάρχει εκταμίευση, αν όχι δεν θα υπάρχει εκταμίευση. Αυτό αλλάζει ε, σε τεράστιο βαθμό τα πράγματα, αυτή η προβλεψιμότητα, να, γνωρίζουμε, να γνωρίζουν και να γνωρίζουμε υπό ποιε συνθήκες θα στείλουμε τη βοήθεια. Στο επόμενο λοιπόν δημοσιονομικό πλαίσιο, να σας πω τι βρίσκω καλό και τι δεν πάει καλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 0,7% στο ε, διαπραγματευτικό κουτί και το θεωρώ καλό. Αλλά υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι κάθε τίτλος γενικός του προπολογισμού πρέπει να υποστεί περικοπές. Και το πακέτο αναπτυξιακής βοήθειας βασίστηκε στο 0,7% και στην βάση αυτήν η Επιτροπή οδηγήθηκε στην κατάρτιση της πρότασης της, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει το 20% της συνολικής βοήθειας. Δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από αυτό τον αριθμό. Θα ήταν άδικο κατά την άποψή μου, γιατί τελικά θα φτάσουμε να υποσχόμαστε άλλα πράγματα και άλλα πράγματα να λέει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν το θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό. Γιατί η αναπτυξιακή, η ε, αναπτυξιακή συνεργασία είναι μια επένδυση για το μέλλον. Είναι μια επένδυση και για το δικό μας μέλλον. Για παράδειγμα, η καταπολέμηση, οδηγεί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι επίσης μια σημαντική οικονομική ευκαιρία. Ευκαιρία για ανάπτυξη. Εάν τα δύο εκατομμύρια νέων. Τα, νέα, δισεκατομμύρια νέων ανθρώπων έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, θα μπορούν να γίνουν και εκείνοι καταναλωτές, θα μπορούν και εκείνοι λοιπόν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό λέω ότι είναι κρίσιμη σημασία να μην βλέπουμε μόνο την ηθική διάσταση, το γεγονό ότι έχουμε ηθική υποχρέωση να βοηθάμε αυτές τις χώρες, αλλά επίσης βλέπουμε και την διάσταση του ότι αυτό είναι μια επένδυση για το μέλλον όλων. Ελπίζω λοιπόν αυτές ε, οι προτάσεις περικοπών να μην ε, συνεχίσουν να εφίστανται στα επόμενα στάδια των διαπραγματεύσεων, γιατί πιστεύω ότι ιδιαίτερα οι ελάχιστα αναπτυγμένες χώρες διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο. Και σήμερα, εάν υπάρχει κίνδυνος σε μία χώρα, αυτό συνιστά κίνδυνο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Νομίζω ότι ε, σας έκανα μια γενική παρουσίαση των κυριότερων ζητημάτων και συμπερασματικά θέλω να πω ότι πάντα με, ε, με ευτυχίζω όταν μπορώ να ανταλλάξω με απόψεις με μια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό με χαρά θα ακούσω τα σχόλιά σας και θα ήθελα να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά. Πρώτον, πρέπει να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε την αναπτυξιακή ατζέντα για μετά το 2015 και αυτό να καταλήξει σε μια γενική παγκόσμια συμφωνία. Όχι απλώς να πούμε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, πρώτον. Και δεύτερον, τα επόμενα 7 χρόνια να δημιουργήσουν μια νέας ποιότητας ε, αναπτυξιακή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η απόφαση σχετικά με την διαφάνεια πρέπει να υιοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα φυσικά και δεν θα αλλάξει τα πράγματα αμέσω. Αλλά είναι μια άλλη νεοτροπία. Και δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε σκέφτονται κάτι παρόμοιο, ίσως όχι από την ίδια αφετηρία, αλλά εάν υιοθετηθεί η Ευρωπαϊκή, ε, ε, υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι τέτοιο, το ίδιο θα κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι μετά θα υπάρχει μια πιο υπεύθυνη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια μεγάλη αγορά, τώρα η Κίνα είναι μια μεγάλη αγορά μου λένε. Ναι, εάν έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να επιβάλλει στην Κίνα να αγοράζει μόνο ε, πρώτες ύλες οι οποίες έχουν παραχθεί νόμιμα. Και επίσης και μια άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ένας νέος αντιπρόεδρος τη Παγκόσμια Τράπεζας για την Αφρική θεωρεί ότι πρέπει να αξιοποιηθούν τα χρήματα που δίνονται σε αφρικανικές χώρες και θεωρεί ότι πρέπει να αξιοποιηθούν για την εξαγωγές αυτών των χωρών. Ναι, υπάρχει το ζήτημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αλλά φυσικά όταν μια επιχείρηση ε, ξεκινά μια διαπραγμάτευση προσπαθεί να έχει ως το δυνατόν μικρότερους ρίσκο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να συζητήσουμε μια σειρά ζητημάτων. Για παράδειγμα, το ζήτημα των αυτόχθονων πληθυσμών. Για παρα... Τα δάση στα οποία αναφερόμαστε θα πρέπει να, έχουν, να υπάρχει νομική προστασία, να, να υπάρχει ε, στη συμφωνία, μια διεθνή νομικά δεσμευτική συμφωνία. Όχι απλώς να λέμε ότι μας ενδιαφέρει το θέμα. η ταχύτητα με την οποία αξιοποιούνται οι φυσικοί πόροι είναι τόσο μεγάλη που θα έλεγα ότι αυτό καθιστά την δράση μας επίγουσα. Γιατί να, ερχόμαστε εδώ στο ζήτημα της βιωσιμότητας. Μπορεί να είναι γρήγορη η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βοηθά και τους πλέον φτωχούς πληθυσμούς και αφού συμφωνήσουμε εμείς πρέπει μετά να συζητήσουμε και με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Κασμάρικ. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε και κύριοι. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Po pierwsze za to, że pan broni MDG, bo rzeczywiście jest e, do 2015 lata i to, że nie osiągniemy wszystkich celów we wszystkich... Έχουμε δύο ακόμη χρόνια μπροστά μας μέχρι το 2015. Και ακόμη και αν δεν πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε τάξει στους αυτούς μας, έχουμε δύο χρόνια μπροστά μας, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούμε να επιταχύνουμε και να σημειώσουμε πιο γρήγορα πρόοδο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί και να τονιστεί ιδιαίτερο. Επίση χαίρομαι που βλέπω ότι ο πλέον σημαντικός στόχος μετά το 2015 θα είναι η κρίζωση της φτώχεια, της ένδυα. Αυτός είναι ένας στόχος που βρίσκεται και κατοχυρώνεται στη συνθήκη και αποτελεί επίση και έναν στόχο ο οποίος επισημαίνεται όλος ιδιαίτερος από, τις, ε, μη κυβερνητικού οργανισμούς. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, χαίρομαι όλος ιδιαίτερος διότι ο Επίτροπος δεν βλέπει έτσι αφηρημένα τους δείκτες και τα με απόλυτα στοιχεία. Θα πρέπει να μπορούμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων με τη βοήθειά μα, Αλλά όλοι αυτοί οι δείκτες πολλές φορές θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε λάθος δρόμο. Να μην μας δείχνουν δηλαδή πώς έχει πραγματικά η κατάσταση. να είναι καλοί οι δείκτες αλλά να μην μπορούν να υλοποιηθούν. Διότι στην Πολωνία έχουμε θαυμάσιους δείκτες για τη στρατηγική μας για το 2020 και για τις επιδόσεις μας. Αλλά παρόλο που οι δείκτες αυτοί είναι τόσο καλοί, ευελιξία φερμή στην αγορά εργασίας ή χαμηλή ανεργία, όλοι αυτοί οι στόχοι δεν έχουν υλοποιηθεί παρόλο που στο χαρτί θεωρητικός είναι εξαιρετική και φαίνονται εξαιρετικοί αυτοί οι στόχοι. Γι' αυτό χαίρομαι που βλέπω ότι κάνει διαφοροποίηση μεταξύ δικτών και της πραγματικής κατάστασης. Να σας ευχηθώ ότι το καλύτερο στη δύσκολη αυτή προσπάθεια την οποία έχετε ξεκινήσει και έχετε αναλάβει, διότι είμαι βέβαιος ότι στα Ηνωμένα Έθνη ο κύριος Μπάνκι Μούν μετά το 2015 έχει αφήσει ανοιχτά τα πράγματα, ανοιχτή την κατάσταση. Και υπάρχει αυτή και η Task Force η οποία θα δει τα πράγματα και μετά το 2015, τη μετά το 2015 εποχή. Και αυτό που βλέπουμε, κοιτάζοντας την κοινωνία των πολιτών, ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα με όλους αυτούς τους στόχους, τους αρνησιακούς στόχους της χιλιετίας. Θα πρέπει κάποιος να καθορίσει προτεραιότητες. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τα πάντα δηλαδή διότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Και το πάνελ στο οποίο είσαστε μέλος εσείς θα πρέπει να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο, το δυσχερές έργο και καθήκον. Και έχω μια ερώτηση που αφορά στη διαδικασία διαβουλεύσεων, αν μου επιτρέπετε τώρα, και που θα ήθελα να σας θέσω. Για σε σχέση με τις επιθυμίες της κοινωνίας των πολιτών μια συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις αρκετά δύσκολες, κοινός εισηγητής Φερρυπίν στα Ηνωμένα Έθνη. Αντιλαμβανόμεθα πόσο δύσκολο είναι να σημειώσει κανείς τέτοια πρόοδο, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βεβαίως θέλουμε περισσότερη συνοχή και συνεκτικότητα στην αναπτυξιακή μας πολιτική, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά πιστεύετε κι εσείς ότι είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος. Υπάρχουν κάποιες κοινέ πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη είναι προβληματικές αυτές. Μπορούμε συνεπώς όλα αυτά τα πράγματα να τα πετύχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ πάντως για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη, λέει ο κύριος Κοντές ε, Λάστρα. Θα ήθελα να σας πω ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι στόχοι της χιλιετίας, αλλά εκπνέουν το 2015 και μέχρι τότε υπάρχουν μεγάλα διεθνή ραντεβού και θα πρέπει να θέσουν τα θεμέλια για τις δεσμεύσεις και τους στόχους που θέλει να βάλει ε, ο κόσμος κατά της ε, φτώχειας. Έχει αλλάξει ο κόσμος και έχει αλλάξει η φτώχεια, το είπατε και εσείς ο ίδιο ε, και εσείς Πρόεδρε. Ε, το 1 δισεκατομμύριο των πιο φτωχών δεν ζουν αποκλειστικά σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, αλλά και μεσαίου πλέον. Γι' αυτό ε, είναι ευθύνη και των κρατών αυτών να θέσουν ε, σε ισχύ και να δρομολογήσουν εκείνες τις διαδικασίες που χρειάζονται για την αναδιανομή του πλούτου και την κοινωνική προστασία, την προστασία της υγείας και τη μείωση συνεπώς των ανισοτήτων. Ποια είναι η κριτική, ότι είναι περιοριστική η στόχη στην εικόνα που δίνουν για την ανάπτυξη και ε, ξεχνούν θέματα ε, όπως είναι η καλή διακυβέρνηση, η ειρήνη, η ασφάλεια, η προστασία των πιο ευαλώτων. Είναι πολλές οι πτυχές ε, της ανάπτυξης που δεν ε, περιλαμβάνονται, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η οικονομική ανάπτυξη. Και αν συμπεριλαμβάνονται, ε, γίνεται με τρόπο ελλειπή. Ας πούμε, η ποιότητα της ελευθερίας και η ισότητα των φύλων. Η δική μου πολιτική ομάδα θεωρεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για το 2015 αυτές τις κριτικές. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, φτάσουμε στο 0,7% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθεια μέχρι το 2015. Είναι νέες οι προκλήσεις, οικονομική, επισητιστική, περιβαλλοντική κρίση. Χρειάζεται να βελτιωθεί η κοινωνική ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα. Με την εκρίζωση της φτώχειας από τις χώρες μας ε, και από τις χώρες γενικότερα πιο συντονισμένα θα πρέπει να απαντήσουμε και χωρίς ε, πρόφαση ε, την να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση και να μην είναι πρόφαση λοιπόν αυτή ε, για να την πληρώσουν πάλι τα 200 εκατομμύρια που ζουν με λιγότερο από ένα ευρώ την ημέρα. Υπάρχουν ε, σαφείς ε, στόχοι μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί. Γνωρίζετε κύριε Επίτροπη ότι σας υποστηρίζει η ομάδα μου για να πάτε στη Νέα Υόρκη με ένα φύλλο πορείας, ένα οδικό χάρτη σοβαρό και ρεαλιστικό για να υπάρχει ένα πλαίσιο ανάπτυξης με οικονομική ανάπτυξη και προσοχή. Ε, μπορεί να φαίνεται χαμηλό το επίπεδο φιλοδοξίας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να βρεθεί η παγκόσμια εκείνη η συμφωνία που θα είναι πιο αποτελεσματική για να ε, ε, τονωθεί η ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σπάνια έχω ακούσει τέτοια εμπνευσμένη ομιλία ε, και τέτοιο ενθουσιασμό από τον Επίτροπο. Το ζούμε, το βλέπουμε ακούγοντά τον. Και λέω τον Επίτροπό μας διότι το θεωρούμε λίγο μέρος της οικογένειάς μας. Και αυτό μου επιτρέπει τώρα να ε, μπω σε θέματα που θα πω με μεγάλη ειλικρίνεια, όπως άλλωστε συζητούν οι οικογένειες. Δεν έχω ε, μεγάλη εκτίμηση, δεν μου αρέσουν τα αριθμητικά στοιχεία, γιατί αυτό δείχνει μια ε, προσέγγιση που θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ε, βεβαίως χρειάζεται πάντα η αξιολόγηση με αριθμητικά στοιχεία. Αυτό που με ενδιαφέρει ένα περισσότερο είναι η μέθοδος. Θεώρησα πάρα πολύ πρωτότυπες τις προτάσεις του κυρίου Πίμπαλξ για το προβληματισμό στην ομάδα εργασίας, στο πάνελ που συμμετέχει. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω να έχουμε μια κοινή ανάγνωση της κατάστασης. Τι εννοώ, ε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να κάνουν μια ανάλυση της κατάστασης και για να το πω σχηματικά, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ανάλυση και μια επισκόπηση και των αποτυχιών αλλά και των επιτυχιών. Παράλληλα, για να ε, γνωρίζουμε από πού κινούμε, ποια είναι η εφετηρία. Η μεγαλύτερη αποτυχία, θα έλεγα, είναι η αδυναμία μια σειρά κρατών να έχουν εκείνη τη διακυβέρνηση που κινουμε ποια ειναι η η μεγαλυτερη αποτυχια θα ελεγα ειναι η αδυναμια μια σειρα κρατων να εχουν εκεινη τη διακυβερνηση που χρειαζεται για να τερματιστεί η διαφθορά, για να μπορεί το κράτος να λειτουργεί και να έχει τις βασικές αρμοδιότητες και εξουσίες του κράτους. Αυτό είναι από τα μεγάλα εμπόδια ε, για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Στις επιτυχίες έρχομαι τώρα. Ας έχουμε λοιπόν το θάρρος να τις πούμε με το όνομά της. Μια πολύ μεγάλη επιτυχής υπόθεση κατά την άποψή μου ήταν η δημιουργία ε, του Παγκόσμιου Ταμείου για την καταπολέμηση του AIDS, ε, της φυματίωσης και της ελονοσίας με μια ανάλυση πάρα πολύ αντικειμενική οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι τα ε, φάρμακα μειώθηκαν στις τιμές του πολλές φορές ε, ε, και 150 φορές φθηνότερα είναι σήμερα για την πρόσβαση σε αντιρετροϊκά φάρμακα για το AIDS. Τώρα, στο μέλλον τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε αυτές τις προκαταλήψεις και τις έμονες ιδέες. Ε, να σταματήσουμε λέμε ότι το εμπόριο καταπολεμά τη φτώχεια. Αυτό είναι η μισή αλήθεια και η μισή αλήθεια είναι και μισό ψέμα. Ε, το εμπόριο μπορεί να είναι ένα μέσο, αλλά αν χρησιμοποιείται με λάθος τρόπο δεν βοηθάει, γιατί μένουν αποκλεισμένοι εκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπων. Γιατί τα λέω αυτά. Ο προλαλής σας σοσιαλιστής συντονιστής αναφέρθηκε σε αυτό, στη διαφοροποίηση δηλαδή. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα τι είναι ε, αυτό που εμπίπτει στη διεθνή αλληλεγγύη και τι εμπίπτει στην εσωτερική εγχώρια αλληλεγγύη. Και εκεί έχει αλλάξει πρόσωπο η φτώχεια. Υπάρχουν πολλοί φτωχοί που δεν έχουν σχέση με τη διεθνή αλληλεγγύη, διότι οι χώρες τους είναι οικονομικά σε θέση να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια τους και δεν ανήκει πλέον στην αναπτυξιακή βοήθεια, ε, δηλαδή των βιομηχανικών κρατών προς άλλα κράτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει και εμείς να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Το λέγουμε και είμαστε και σχεδόν ομόφανοι σε αυτό, αλλά όταν πρόκειται να ψηφίσουμε τα κείμενα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά πλειοψηφία καταψηφίζουμε και αντιφάσκουμε. Ας εμπνευστούμε από τα ίδια μας τα λόγια και όχι από τα έργα μας. Λοιπόν, θα χρειαστεί να οριστεί η ευθύνη του καθενός. Εγώ δεν δέχομαι πλέον να κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτος δωρητής ότι είναι λέει υπεύθυνη για την αύξηση του αριθμού των φτωχών στις αναδυόμενες χώρες που κατά τα άλλα έχουν αρκετά λεφτά για να αντιμετωπίζουν την ίδια τους τη φτώχεια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πραγματικά ε, ανυποχώρητοι και ε, ας μας θεωρήσουν ότι τους ε, χαλάμε εκεί ε, στο πάνελ την υπόθεση. Εντάξει, οι στόχοι της χιλιετής με την παλιά ή τη νέα τους εκδοχή, αλλά θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να θέτουμε και αυτά τα θέματα επιτάπητος για τις συζητήσεις. Και βέβαια είναι πρόβλημα το 0,7% της αναπτυξιακής βοήθειας. Και εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Είναι μια αποτυχία, τη φοβάμαι, δεν την αποκλείω, ούτε την επιθυμώ. Αλλά ε, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα μέσα εκτός εκείνων που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις και η απόλυτη ένδυα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στη συνείδηση όλων εκείνων που ε, φέρουν την ευθύνη, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και κατά κύριο λόγο αυτούς που κρύβονται πίσω από ε, το πρόσχημα της ε, εθνικής κυριαρχίας για να μην καταπολεμήσουν τη φτώχεια στη χώρα τους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Έχω δύο σημεία να μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο είναι η έλλειψη συνεργασίας και ε, ο πάρα πολύ επιλεκτικός τρόπος με τον οποίο η ΜΚΟ ε, αρνούνται συμμετοχή ευρωβουλευτών σε διασκέψεις που διοργανώνονται με χρήματα των φορολογουμένων. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας και για την πρόταση για ενισχυμένη συνεργασία. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και να σας πω πώς μια ευρωπαϊκή ΜΚΟ συμπεριφέρεται σε ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Euro NGO είναι ο φορέας που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φτάσουμε στους στόχους της ηλιετίας για την ε, υγεία των μητέρων, την αναπαραγωγική και ε, γενετήσια υγεία. Και εργάζονται πάρα πολύ στενά σε συνεργασία με ε, τις δικές σας υπηρεσίες. Τούτη την Πέμπτη διοργανώνουν μια διεθνή διάσκεψη για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία στις Βρυξέλλες για να ορίσουν την ατζέντα για μετά το 2015. Κυριολεκτικά όλες οι ΜΚΟ της Ένωσης είναι προσκεκλημένες και όλες οι αρμόδιες και όλοι οι φορείς. Εγώ ζήτησα επίσημα να προσκληθώ ως ε, ε μέλος της Επιτροπής ΔΕΒΕ που ανησυχώ για αυτά τα θέματα και με τρόπο πάρα πολύ αγενή μου απήντησε η Euro NGO και μάλιστα η Άν Σβένσον, πρόεδρος, μου είπε ότι δεν χρειαζόμαστε, λέει, τη, βοήθειά της και μάλιστα το τύπωσα γιατί είναι απίστευτο αυτό που μου λέγουν. Η γενική μας διεύθυνση χρηματοδοτεί, η δική σας ε, χρηματοδοτεί αυτή τη Euro-NGO και η κυρία Φρανσουάς Μωρό εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη διάσκεψη, πάλι της δικής σας γενικής διεύθυνσης. Αλλά τα μέλη της δικής μας Επιτροπής Ανάπτυξης αποκλείονται από μια διεθνή διάσκεψη που αντιμετωπίζει τα ίδια θέματα με τα οποία σήμερα εσείς σας ασχολείστε. Γνωρίζω ότι εσείς δεν ε, διοργανώνετε αυτές τις ε, διασκέψεις Βρυξέλλες για τη Euro NGO. Παρόλα αυτά είναι το βασικό εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πληρεί τους στόχους αυτούς και ε, το θέμα 5, το, το στόχο υπαριθμών 5 για την υγεία των μητέρων και την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία των γυναικών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο αφορά τις κατευθυντήριες αρχές για την καταπολέμηση της απόλυτης ένδυας και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει υποβάλει ο ειδικό εισηγητής για την απόλυτη ένδυα και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στο Συμβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από λίγες εβδομάδες. Στο σημείο 72 τονίζεται η αρχή ε, της γονικής ευθύνης ε, σε ό,τι αφορά τη φτώχεια των παιδιών. Και ρωτώ, πώς σέβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση την αρχή της γονικής ευθύνης σε αυτό το θέμα της παιδικής φτώχειας. Η παιδική φτώχεια είναι ένα θέμα ε, πάγιο και διαρκές, αλλά τι δουλειά έχει η γονική ευθύνη και πώς ε, ε, ενέχεται αυτή συγκεκριμένα. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Πίμπαλξ για να απαντήσει σε αυτή την πρώτη ομοβροντία ερωτήσεων. Well, thank you very much. Ευχαριστώ όλους σας για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας και το προσωπικό μου ακούει και σας ακούει. Επομένω, οι υποδείξει σα, οι προτάσει σα έχουν κρίσιμη σημασία για μα και στο πώ αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά και πώ θα τα αντιμετωπίσουμε, διότι θέλουμε να είμαστε έτοιμοι προκειμένου να ετοιμάσουμε μια ανακοίνωση προ υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρί του χρόνου. Νομίζω λοιπόν πω έχει κρίσιμη σημασία να γνωρίζουμε την άποψή σα. Τώρα, όσον αφορά κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία τέθησαν, ο Φίλιπ ρώτησε για τον νέο εισηγητή. Εγώ πάντοτε επιδεικνύω σκεπτικισμό όταν μιλάτε δηλαδή για τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού οργάνου. Τώρα βεβαίως όλα δεν τα γνωρίζω και για μένα είναι ένας κρίσιμος εταίρος. Η UNDP νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή θέση για να εργαστεί σε θέματα σαν και αυτά. Νομίζω ότι ο βασικός μετέρος είναι η UNDP για μένα. Και βεβαίως ενδεχομένως να μην έχουν επαρκείς πόρους, αλλά αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή γιατί τα Ηνωμένα Έθνη θα αποφασίσουν μόνα τους το τι θέλουν. Αλλά νομίζω πως η UNDP βρίσκεται σε καλή θέση. Διότι έχουν αφιερώσει και χρόνο στο ζήτημα αυτό και τα νέα θεσμικά όργανα πάντα δημιουργούν πρόβλημα χρηματοδότησης και συνεκτικότητας και συνοχής με άλλα. Επομένως νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πρόκληση και μιλήσατε για την βιώσιμη ενέργεια για όλους του Υπάρχει ένας ειδικό απεσταλμένος και CEO και θα θέλαμε να το υποστηρίξουμε, αλλά δεν υπάρχει μια οργάνωση η οποία θα μπορούσε να, αναλάβει αυτός για να ξεκινήσει την, αυτή την διεργασία. Νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν και πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Αν δοθούν, να θέλετε, και απαραίτητοι πόροι και αναντηθούν αυτά τα καθήκοντα σε υφιστάμενου φορεί. Τώρα, για τα 2015 και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε για τη διαφοροποίηση, θα συνεχίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να παίζουν τον ρόλο μας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παγκόσμιος παίκτη. Μέσω περιφερειακών προγραμμάτων και θεματικών προγραμμάτων θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε. Διότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κρίσιμος σε αυτόν τον πολυμερή κόσμο, διότι προϊόντος του χρόνου νομίζω ότι έχει παρέλθει η εποχή και ο καιρός, αν θέλετε, των υπερδυνάμεων. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολυμερής πλέον και πρέπει να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες μας προκειμένου να βρούμε τις καλύτερες και τις πιο συμφέρουσες δυνατότητες και ευκαιρίες για όλους. Και όταν ο Τσάρλς μίλησε προηγουμένως, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ενθάρρυνση για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ξέρω ότι δεν είμαστε τέλειοι Πόρο απέχουμε τη τελειότητα, Αλλά ό,τι κάνουμε ε, ε, γίνεται σεβαστό. Γίνεται σεβαστό παντού. Και ακόμη δηλαδή που έχουν ασκήσει κριτική, σέβονται αυτό το οποίο κάνουμε. Και αυτό νομίζω μας προσφέρει αν θέλετε μια κάποια ικανοποίηση γνωρίζοντας ότι γίνεται σεβαστή η προσπάθειά μας αλλά και αποτελεί και μια πρόκληση συνεχώς. Ο Τσάλς είπε πολλά σε παγκόσμιο επίπεδο νομίζω είχαμε τεράστια επιτυχία. Γιατί κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι μιλούσαμε δηλαδή για το, ότι, για το AIDS και δεν έχει εξαφανιστεί βεβαίως. Παραμένει ζήτημα το AIDS και η αντιμετώπιση του. Αλλά νομίζω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται η προσπάθεια και θα μπορέσουμε αν θέλετε να εκριζώσουμε, να εξαλείψουμε δηλαδή το, το βασικό αίτιο του AIDS, Ερπίν. Εστιάζοντα την προσοχή μα πάνω σε ορισμένα θέματα, πολλά μπορεί να πετύχει κανεί. Αλλά πιστεύω επίση ότι υπάρχει ένα περιορισμό σε σχέση δηλαδή με το τι μπορούμε να επαναλάβουμε εμεί. Διότι η ισχύ μα είναι να εστιάσουμε την προσοχή μα δηλαδή σε τρει βασικέ ασθένειε και νόσου. AIDS, HIV, ελαιονισία και φυματίωση και νομίζω ότι πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αυτό για να καταπολεμήσουμε τις ασθένειες αυτές. Και μιλώ, μιλούμε επίσης και για, τη, για τα εμβόλια και για την... Ε, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος δεν είναι ακόμη ενωμένο, γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν χώρες κράτη. Θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε και να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ μια εθνική προσέγγιση και μια θεματική προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε και χρειάζεται. Δεν λέμε δηλαδή τα δικά μα χρήματα είναι καλύτερα από τα χρήματα κάποιου άλλου. Αλλά εκεί όπου βλέπουμε και τα θέματα είναι πολύ συγκεκριμένα, σαφώ ορισμένα. Α υιοθετήσουμε αυτή τη θεματική προσέγγιση, διότι νομίζουμε ότι αυτή είναι και η πιο αποτελεσματική. Αλλά δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε. Διότι για κάποιες χώρες, σε κάποιε χώρε υπάρχει διαφθορά, υπάρχουν προβλήματα. Γιατί σε τελική ανάλυση Εργαζόμαστε με τους λαούς των χωρών αυτών. Και πιστεύουμε δηλαδή ότι οι χώρες αυτές θα ξαναβρεθούν στο σωστό δρόμο. Γιατί δεν υπάρχει στόχη υπάρχουν κάποιοι κυβερνητικοί δείκτες. Άρα τουλάχιστον και σύμφωνα με τη δική μου την εμπειρία θα έλεγα ότι οι χώρες αυτές βελτιώνουν την κατάστασή τους. Και πολλές φορές ασκούμε κριτική και τις στιγματίζουμε, διότι δεν είναι τέλειες χώρες. Αλλά πρέπει επίσης να δούμε και την πρόοδο που σημειώνεται στις χώρες αυτές και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες. Γιατί μίλησατε προηγουμένω για την ε, Λιβερία. Όντως, η διαδικασία αδειοδότησης δεν είναι και τόσο διαφανής. αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι η κυβέρνηση σταμάτησε τη διαδικασία αυτή και έκανε και την πρώτη της επανεξέταση. Και τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται και μια δεύτερη επανεξέταση της καταστάσεως αυτής ήταν σημαντικό ότι η κυβέρνηση της Λιβερίας αντίδρασε όχι δηλαδή μετά από δική μα πίεση αλλά από πίεση τη κοινωνία των πολιτών τη. Και αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία στηρίζουμε. Βεβαίω δεν ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία όσοι θα ελπίζαμε, αλλά πιστεύουμε ότι κινείται προ την ορθή κατεύθυνση και νομίζω ότι θα βρούμε πολλέ χώρε του κόσμου στι οποίε γίνεται αυτό. Θα πρέπει συνεπώ να ενθαρρυνθούμε και να παροτρύνουμε και να ενθαρρύνουμε όσον αφορά το εμπόριο τώρα. Πράγματι, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει και πάρα πολύ το εμπόριο. Νομίζω ότι ένα βιβλίο που γράφει σχετικά με το θέμα αυτό δεν το προσεγγίζει σωστά. Το εμπόριο έχει αντίκτυπο, έχει επίπτωση. Αλλά δεν βγάζει στις χώρες δηλαδή και το λαό από τη φτώχεια τους με το εμπόριο. Απλώς ε, κάνει του πλούσιους πλουσιότερους αξιοποιώντα τα εθνικούς πόρους αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού αυτού δεν είναι πλούσιο, είναι πτωχό. Επομένως νομίζω ότι μας ξαναφέρνει στον δρόμο. Διότι αν πάρεις σε οδήποτε αφρικανική χώρα, σαν παράδειγμα, οι υποδομές είναι ένας τρόπος, δηλαδή πώς θα βοηθήσουμε δηλαδή, τους φτωχούς και θα τους ε, βελτιώσουμε την οικονομική τους κατάσταση. Επομένως νομίζω πως έχει κρίσιμα σημασία αυτό που ξεκινήσαμε με τη διαφάνεια νομίζω πως η... στόχος μας θα πρέπει να είναι η διαφάνεια. Δηλαδή να φύγει κανείς με τα χρήματα στην τσέπη του αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Και αυτό είναι, θα είναι δικό μας λάθος, δεν είναι λάθος αυτών των φτωχών χωρών. Διότι ζουν, αν θέλετε, κάτω από παγκόσμιε συνθήκε και δεν πιστεύουν οι χώρε αυτέ στο μέλλον του. Και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και όσο το κρατήσουμε αυτό για τον, για τον λόγο, τότε δεν μπορέσουμε ποτέ να κερδίσουμε την μάχη αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να στηρίξουμε τις ε, χώρες αυτές, να στηρίξουμε τη δημιουργία βιώσιμων οικονομιών και επιδεικνύοντας διαφάνεια. Και εμείς αλλά και εκεί. Να δεχόμαστε δηλαδή στη δική μας τις αγορές εδώ πέρα κάτω μόνο νόμιμα προϊόντα και βεβαίω ε, να φροντίσουμε ότι οι χώρες αυτές, οι τρίτε χώρες δηλαδή, να έχουν μια πολύ καλή, μια ορθή δηλαδή και χρηστή διαχείριση της παραγωγή του. Νομίζω πω αυτό είναι ένας δρόμος τον οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσουμε γιατί είναι πάρα πολύ καλός και θα μας βοηθήσει. Λυπούμε, αν θέλετε, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, κλονίστηκα μάλλον από αυτά που είπε η κυρία Ζαμπόρσκα. Το μοναδικό πράγμα θα μπορούσα να πω, ότι θα γράψω μια, ένα γράμμα στην ε, οργάνωση στην οποία αναφερθήκατε. Εμείς απλώς τη στηρίζουμε, δεν είμαστε μέτοχοι της ούτως είπεν. Αλλά πραγματικά κλονίστηκα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ποτέ. Διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προφανώς πρέπει να μπορεί να συμμετέχει. Είναι ο, ο πλέον ζηλευτός, αν θέλετε, τέλος. Αν σας λένε όμως δεν σας θέλουμε, αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται σεβαστή και δεν τηρείται, τηρούνται οι δημοκρατικές διαδικασίες. Θα γράψω εγώ και θα ζητήσω εξηγήσει από αυτόν τον Ευρωπαϊκό Μίκιο. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάτι το οποίο οργανώνει και οργανώνει τα του μη κυβερνητικού οργανισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη στηρίζουμε απλώ. Αλλά νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα και μπορούμε να ζητήσουμε εξηγήσει. Έτσι νομίζω απαντώ στο ερώτημα σα. Όσον αφορά τώρα την γονική ευθύνη. Είναι περίπλοκο το όλο ζήτημα και δεν εργαζόμαστε πολύ προ την κατεύθυνση αυτή. Καταλαβαίνω τι λέτε μεν, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με την ε, πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Νότια Αφρική επισκέφτηκα ένα έργο. Απλώς το συγχρηματοδοτούσαμε. Ένα γερμανικό έργο. Και έχει σχέση με το ποδόσφαιρο δηλαδή. Δηλαδή οργανώνει ποδοσφαιρικού αγώνε και τέτοια πράγματα, αλλά κατά τη διάρκεια αυτών να μπορέσει να εξηγήσει πολλά πράγματα. Αλλά ε, οι πατεράδε δεν ήταν ποτέ εκεί. Το πρόβλημα αυτό είναι βαθιά ριζωμένο στη χώρα αυτή. Όχι που δεν ε, αρέσει στους πατεράδες δηλαδή, αλλά η μητέρα είναι που έχει αναλάβει και αναλαμβάνει την ευθύνη των παιδιών, γιατί αυτή θα πρέπει να τα θρέψει. Επομένως πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Γιατί εκεί υπάρχει ακόμη apartheid, έτσι τουλάχιστον το αποκαλώ εγώ στην Νότια Αφρική. Και νομίζω ότι η κοινωνία μας, αν θέλετε, ακόμη φέρνει τα τραύματα, αν θέλετε, από του παρελθόντος στην πλάτη της. Υπάρχουν πολλές καλές οικογένειες, αλλά υπάρχουν κάποια βαθιά ριζωμένα προβλήματα, τα οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Να στηρίξουμε πραγματικά τα παιδιά. Γιατί και αυτά θα φτιάξουν οικογένειες και έτσι οι οικογένειες του θα είναι πολύ πιο ευτυχισμένες από ότι είναι οι τωρινέ τους οικογένειες οι σημερινές του οικογένειε και θα πρέπει εδώ να προσφέρουμε δηλαδή τι βασικέ υπηρεσίε παιδεία. Γιατί μόνο έτσι θα έχουν περισσότερες ευκαιρίε και πιθανότητε να πετύχουν και να μπορέσουν να καταλάβουν επίσης και τις αξίες τη ζωής. Όπως επίσης και να δώσουμε και να εξασφαλίσουμε και ένα κατάλληλο σύστημα κατοικιών. Στέγης δηλαδή. Γιατί πολλοί φερρυπίν ε, γονείς έχουν πεθάνει λόγω AIDS και τα παιδιά αυτά ζουν, αν θέλετε, χωρίς γονείς και προσπαθούν να επιβιώσουν. Είναι περίπλοκο το ζήτημα αυτό, είναι από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου και είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουμε και να ενισχύσουμε τις κυβερνήσεις και τις προσπάθειες που καταβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις όμως το αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά το ζήτημα. Έχουν γίνει βέβαια κάποιες προσπάθειες αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα. ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριου Νόησαρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πολλές φιλοφρονήσεις ακούσατε και επένους και δικαίως. Νομίζω ότι στο πρόσωπό σας η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προετοιμασία α, της νέας εποχής είναι σε καλά χέρια. Όχι μόνο επειδή είστε επίτροπος, αλλά επειδή είστε και ο συγκεκριμένος επίτροπος με την προσωπικότητά σας. Εγώ θα επικεντρωθώ στην καταπολέμηση της φτώχειας, που είναι και ο μεγάλος στόχος και εξακολουθεί να παραμένει από τους στόχους της χιλιετίας. Αλλά στην καταπολέμηση της φτώχειας παγκοσμίω έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και τα διαρθρωτικά σημεία της ανισότητας στη φτώχεια και η έλλειψη της περιβαλλοντικής εφορίας είναι κάποιοι ε, στόχοι, κάποιες πτυχές που έχουν παραγωνιστεί. Ε, ε, είπαν και άλλοι συνάδελφοι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τακτική για την καταπολέμηση της στόχιας. Το 1990 το 93% των πιο φτωχών ήταν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2008 το 72% των πιο φτωχών ζουν σε χώρες με εσέου εισοδήματος. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει και εκεί να αλλάξουμε και στρατηγική. Και στους στόχους της χιλιετίας, όσο και αν τους υπερασπίζομαι και όσες επιτυχίες και να έχουμε, ε, υπάρχουν μερικά φαινόμενα που ανέφερε και ο Ρικάρδο, τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη. Ανθρώπινα δικαιώματα, συμμετοχή του κόσμου, κράτος δικαίου, ε, ε, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη στη διανομή. Και για τη νέα εποχή, μετά το 2015, χρειαζόμαστε μια νέα φιλοσοφία. Κατά την άποψή μου, μέχρι σήμερα οι στόχοι της χιλιετίας είναι κάτι που έχει επιβληθεί από πάνω προς τα κάτω, από το βορρά στο νότο και ο 8 στόχος, Φερρυπίν, που είναι η παγκόσμια εταιρική σχέση, δεν έπιασε πάρα πολύ. Ε, και θα πρέπει περισσότερο να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Έχουμε καλές οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, έχουμε καλές ΜΚΟ, αλλά αυτά ε, υπάρχουν στο βορρά στην Ευρώπη και δεν επαρκούν και έχουμε και μια καταναλωτική συμπεριφορά, έχουμε τρόπο παραγωγή σε, σε βιομηχανικέ χώρε, συγγνώμη, έχουμε εμπορικέ συμφωνίε στην κοινή γεωργική πολιτική και θέματα εξαγωγών όπλων που πρέπει να τα ξαναδούμε. Και ε, πέρα από ε, τον 8ο στόχο για τη μελλοντική οριοθέτηση των νέων στόχων θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Και τελευταίος. Κλείνει το μικρόφωνο, πρόεδρος, και δεν ακούμε σε ποιον... Α, ο κύριος Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ. Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω για τα νοσήματα, αλλά τα είπατε μόνο σας. Ε, να σας ρωτήσω κάτι για το καθαρό νερό, το πόσιμο νερό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέσσερα μέλη πήγαμε στην Ινδία, νομίζω το Μάρτι φέτος, για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια απάντηση, αν πρέπει να βοηθήσουμε την Ινδία ή όχι και ένα τμήμα της επίσκεψης ήταν ε, στο Ρατζαστάν, στην έρημο, σε ε, μια εγκατάσταση επεξεργασίας υδάτων που έχουμε εμείς χρηματοδοτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την έρημο βγάζανε νερό, χειρονακτική εργασία. Βέβαια, οι πλούσιοι στο Νέο Δελχή δεν ε, δέχονται, δεν τους αρέσει να τους δίνει λεφτά η Ευρώπη, αλλά τα 500 εκατομμύρια των φτωχών Ινδών χρειάζονται ε, πραγματικά ε, πολύ έντονα τη βοήθειά μας. και ήταν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που μας έκανε και ήθελα να μιλήσω λοιπόν για το πόσιμο νερό και τις αρρώστιες, αλλά τα είπατε μόνο σας. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Έχετε παρακαλώ το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις και να ολοκληρώνετε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρα. Θα αρχίσω με την ερώτηση του κυρίου Νόισερ για την σημερινή κατάσταση και τις προοπτικές. Ε, υπάρχουν διάφοροι πυρογνώμονες που λέγουν διάφορα στοιχεία, αλλά εγώ νομίζω ότι θα αλλάξει η παγκόσμια φτώχεια θα μειωθεί σε χώρες μεσαίου εισοδήματος με γρήγορο ε, τρόπο, ενώ στις πιο φτωχές χώρες του χαμηλού εισοδήματος, επειδή αυξάνεται με τεράστιες ε, ταχύτητες και ρυθμούς ο πληθυσμός τους, θα αυξηθεί. Και αλλού, και δεν είναι δική μου ηρολογία αυτή, σε εύθραυστα ε, και αποτυχημένα κράτη μεσαίου εισοδήματος. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου εφευρέσεως. Και υπάρχουν τέτοιες χώρες. Αναφέρω δύο το Πακιστάν και η Νιγηρία. Ε, τεχνικά είναι μεσαίου εισοδήματο, αλλά ξέρουμε πόσο εύθραυστη ε, ε, είναι η κατάσταση εκεί και εκεί υπάρχει το θέμα αυτό, το ρίσκο της φτώχεια. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση, αλλά δεν είναι μόνο οι λιγότερο ανεπτυγμένες, αλλά είναι και ευαίσθητες χώρες, οι εύθραυστες και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε με προστιθέμενη αξία και εκ των προτέρων. Τι περιμένω από το παγκόσμιο πλαίσιο, να αναγνωρίσει τις ε, ε, προσπάθειες που κάνουν η Κίνα και η Ινδία και μάλιστα να τους βάλουμε και υποχρεώσεις ε, να συνεργαστούν για να κρυζώσουν τη φτώχεια στις δικές τους χώρες. Το είπε και ο κύριος Νιούτον Ντάν. Στην Ινδία υπάρχουν πολύ μεγάλοι θύλακες φτώχειας, αλλά δεν θέλει η Ινδική κυβέρνηση να εργαστεί ε, μαζί μας για αυτό το θέμα, στο να λάβουν οι ίδιοι όμως, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γιατί είναι δίκαιο και θα αναγνωριστεί, ακόμα και αν μειωθεί η φτώχεια ε, στην Κίνα και στην Ινδία. Είναι τεράστια η προσπάθεια και το έργο αυτό, αλλά η δική μας βοήθεια δεν έχει μεγάλο νόημα εκεί. Ας πούμε μια χώρα όπως είναι το Νεπάλ, από πιο ε, φτωχές χώρες και λιγότερο ανεπτυγμένες και κάνει πρόοδος, η δικιά μας βοήθεια ε, πιάνει μεγάλο τόπο στο Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς ε, θα μπορούσε να κρυζωθεί η φτώχεια αν δεν υπήρχαμε εμείς. Δεν μπορώ καν να το διανοηθώ. Και αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε, ε, επιμένουμε σε αυτό. Τώρα ο κίνδυνος για την άνωθεν ή ε, κάτωθεν προσέγγιση. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικές οι πραγματικότητες. Εγώ αυτό που βλέπω στη δουλειά μου είναι ένα χάσμα, έτσι, μια διαίρεση βορανότου δεν ξέρω από πού προέρχεται, μάλλον ανάγεται σε πολύ παλιούς καιρούς, ε, ότι ο Βορράς είναι οι χώρες του ΩΣΑ ε, και ο Νότος είναι αναπτυσσόμενες, οι 77 κτλ. Αυτό δεν ισχύει γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα στο Βορρά. Υπάρχει η Λετωνία ας πούμε που θα μπορούσε να θεωρηθεί κάπως διαφορετικά και αν είχαμε επιλέξει άλλο τρόπο ζωής θα ήμασταν χώρα του Νότου, ξέρω εγώ. Όλα αυτά είναι τεχνητά κατά την άποψή μου ως διαχωρισμοί, αλλά υπάρχουν και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε. Και δυστυχώς δεν προχωρούμε όπως θα ανέμενε κανείς. Οι ορισμένοι έχουν δείξει αποτελεσματικότητα με αυτή την διάνοιξη που είναι η Ινδία, η Κίνα και τώρα προετοιμαζόμαστε για την παγκόσμια αυτή εταιρική σχέση για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, νομίζω έτσι επιγράφεται. Στην πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει μέχρι τα τέλη του έτους, κάπου εκεί, η λογική ποια ήταν, η αναπτυξιακή συνεργασία να φύγει από τον ΟΣΑ από την ΤΑΚ που κάνει διάφορες μελέτες και τα λοιπά, αλλά να περάσουμε σε μια νέα δομή, σε μια νέα μορφή. Και αν δείτε ποιο δραστηριοποιείται εκεί, η Νιγηρία, ο Υπουργό Οικονομικός ο της Νιγηρίας, η Ινδονησία και πιστεύω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την προθυμία της Ινδονησίας και να συνεργαστούμε, αλλά οι μεγάλοι, οι μεγάλοι τρεις ας πούμε, Κίνα, Ινδία και Βραζιλία αυτή τη στιγμή διστάζουν. Δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή μπουν. Αλλά το θέμα είναι και ποιος αναπτύσσει αυτή τη φιλοσοφία. Ε, το πρόγραμμα για την ανάπτυξη του ΟΗΕ. Αλλά η νέα αρχιτεκτονική δεν δημιουργείται. Και εγώ τι φοβάμαι. Γιατί είναι και πραγματικότητα. Πρώτον, φοβούμε ότι ο ΣΑ και πάλι ΝΤΑΚ για τα επόμενα 7 έτη θα είναι κινητήρια δύναμη. Και εγώ δεν δέχομαι την ε, ε, τις επικρίσεις ότι οι δωρητές ορίζουν. Όχι, μα έγινε αυτή η κίνηση, ε, αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να καθοδηγεί όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα, όσο και αν δεν μας αρέσει. Και η δεύτερη σκληρή πραγματικότητα είναι οποιοδήποτε και είναι το πλαίσιο που θα δημιουργηθεί για την πρόταση, θα πρέπει αυτό να γίνουν συνενετικά. Τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να πείσουμε τους εταίρους μας αυτή τη φορά, να βρούμε μια καλύτερη φόρμουλα για να αισθάνονται άνετα με τα παγκόσμια ε, φόρα. Δηλαδή, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, όπως καμιά φορά χρειάζεται να εξηγώ, τι σημαίνει πράσινη ανάπτυξη. Και μου λένε και τι είναι η πράσινη ανάπτυξη. Τι είναι, πράσινα άλογα. Η πράσινη ανάπτυξη σημαίνει αηφόρος, βιώσιμη ανάπτυξη που να χρησιμοποιεί όλο το δυναμικό που έχει ο καθένας. Ε, αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Ε, ε, τέτοιο είδους παρεξηγήσεις νομίζω θα πρέπει να τις αποφεύγουμε. για το πόσιμο νερό, το καθαρό νερό και τα υγειονομικά ζητήματα. Βεβαίως, ε, ό,τι έχει να κάνει με τη γεωργία, τα περισσότερα ζητήματα, την επιστηστική ασφάλεια ε, και άλλα τέτοια συναφή και θέματα υγείας έχουν να κάνουν με το καθαρό νερό ε, και τα θέματα τα υγειονομικά. Είναι ένα εγκάρσιο θέμα που καλύπτει πάρα πολλούς τομείς. Το νερό λοιπόν, τα τρόφιμα και η ενέργεια. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις ε, είναι κρίσιμο να έχεις πρόσβαση στην ενέργεια για να καθαρίσεις το νερό ας πούμε ε, ή ε, να έχεις πετρέλαιο για να παράγεις τρόφιμα η ενέργεια. Και το συζητούμε αυτό και με την Ινδία και σε διμερή συνεργασία φαίνεται ότι καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρώνεται σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στις πιο ε, ε, λιγότερο αναπτυγμένε. Και αν θέλουν τα κράτη-μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο, διμερό βεβαίω να συνεργάζονται. Ε, η πρότασή μα καλύπτει μόλι το 12% των δεσμεύσεων άλλωστε. Οπότε έχουμε περίπου 90% για να καλυφθεί αλλού. Λοιπόν, Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταλλαγή αυτή. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και είμαι πρόθυμος ε, να δεχτώ τις προσωπικές ε, προτάσεις των μελών της Επιτροπής σας, τι πρέπει να πάω να πω στο πάνελ και το πάνελ ξέρετε ένα βήμα μόνο είναι. Δεν είναι και αυτός σκοπός. Ε, δίνει στο Γενικό Γραμματέα κάποιες ιδέες. Είναι μακράς πνοής αυτή η υπόθεση. Αλλά είναι σημαντικό το πάνελ να μπει στη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι κρίσιμο. Το πρώτο βήμα να μην είναι στραβό. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που είπε ο Φιλίπ, ότι χρειάζονται προτεραιότητε. Δεν μπορούμε να τα πετύχουμε όλα ταυτόχρονα και ίσω αυτό είναι μεγαλύτερη δυσκολία. Γιατί εύκολο είναι να προτείνει τα πάντα, αλλά όταν προσπαθεί να κόψει από αυτό το ευκολόγιο, ε, είσαι στόχο κριτική ότι δεν έχει αρκετή φιλοδοξία. Ε, κάπου πρέπει έτσι κάπω να τετραγωνίσουμε αυτό τον κύκλο και σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που μοιραστήκατε μαζί μας ε, αυτό το πρωτόλιο στάδιο του διαλόγου για την περίοδο μετά το 2015 και το σημειώσαμε αυτό ότι προσκαλείτε τα μέλη να κάνουν προτάσεις, να σας υποβάλουν ιδέες για το τι θα πρέπει να συζητηθεί στο πάνελ. Νομίζω ότι εξ ονόμα της Επιτροπής, ε, μάλλον τα μέλη της Επιτροπής μας τα άκουσαν αυτά με μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Δεν έχουμε σημεία για τα διάφορα της ημερησίας διάταξης και η επόμενη συνεδρίασή μας θα τελεστεί εδώ στις Βρυξέλλες. Δευτέρα 5 Νοεμβρίου από τις 15 το μεσημέρι μέχρι τις 19.30 και την, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ όλους και όλες σας για την παρουσία και τη συνεργασία τη. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερω του διερμηνείς η Πρόεδρος που έπρεπε να παίξουμε διάφορους γλωσσικούς συνδυασμού και είναι πολύ δύσκολη η οργάνωση τη εργασία εντός των καμπινών της διερμηνία λόγω των κοινών αυτών συνεδριάσεων που είχαμε για το βραβείο Ζαχάροφ. Ευχαριστώ επίσης και τους κλητήρες. γιατί πολλοί κόσμος ήθελε να παρακολουθήσει τη διαδικασία ψηφοφορία μας. Ευχαριστώ λοιπόν σε όλους σας και όλες σας.